Άρχεται λοιπόν η συνεδρίαση, η συντακτική συνεδρίαση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη το στόχο τη ε, σημερινή μα συνάντηση. Είμαστε λοιπόν εδώ για να ε, συγκροτήσουμε το Προεδρείο της Επιτροπής που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους. Και αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό 191 του Κοινοβουλίου θα ακολουθήσουμε την εξή σειρά εκλογής. Πρώτα θα εκλέξουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και κατόπιν θα προχωρήσουμε στην εκλογή των αντιπροέδρων. Θα ήθελα να σα ανακοινώσω ότι διαθέτουμε την απαραίτητη απαρτία που ε, με βάση τον κανονισμό 195 παράγραφος 2 είναι 19 μέλη των τέταρτων. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να υποβάλλετε τις υποψηφιότητες για τη θέση του Προέδρου που μπορεί να γίνει είτε μέσα από μια ε, πολιτική ομάδα είτε από το 5% 31, ε, ε, με βάση τον κανονισμό 13.1. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων να μας καταθέσουν τις προτάσεις. Ο κύριος Αλαφράγκα εκ μέρους του ΕΛΚ. Εξ ονόματος της ε, ομάδας του Λαϊκού, Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και σύμφωνα με τον κύριο Μπροκ, καινούργιο μου σύντροφο, de facto, θα προτείνουμε τον κύριο Αλμπερτίνη. Ε, αντιπρόεδρο της, πρώην αντιπρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών πρώην δήμαρχο του Μιλάνου, έχει μακρά πορεία, έχει συναντήσει πάνω από 40 αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων. Λοιπόν, προτείνουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Αλμπερτίνη. Thank you, uh, Are there any... Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σαλαφράγκα. Άλλος παρακαλώ επιθυμεί κάποιος άλλος να καταθέσει ή να ανακοινώσει υποψηφιότητα. Κανείς άλλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε λοιπόν στον ε, ε, διορισμό του Προέδρου αυτής της Επιτροπής. Ε, επιθυμεί κανείς την μυστική ψηφοφορία. Αυτό, αν το θέλετε, πρέπει να το ζήσουν 13 μέλη με το ενέκτον με βάση τον κανονισμό 191 δεύτερη υποπαράγραφος. Κανείς λοιπόν δεν ζητάει το λόγο. Κατόπιν τούτου ο κύριος Αλμπερτίνη είναι ο μόνος υποψήφιος και ως εκ τούτου ο κύριος Αλμπερτίνη εκλέγεται πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον κύριο Αλμπερτίνη και θα ήθελα να του ζητήσω να έρθει εδώ στο βήμα να λάβει τη θέση του Προέδρου για να προχωρήσουμε στην ε, περαιτέρω εκλογή των ε, υπολείπων των αντιπρόεδρων. Επιτρέψτε μου πριν ε, συνεχίσουμε τις ε, εργασίες μας στα πλαίσια της Επιτροπής μας, να πω δύο λόγια μονάχα για τα όσα συμβαίνουν. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους παρισταμένους συναδέλφους, για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Ιδιαίτερος δε τα μέλη της Ιταλικής Αντιπροσωπείας που με επέλεξαν. Παρόλα όλα αυτά, αισθάνομαι ότι οφείλω να πω δύο λόγια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου απέναντι σε ένα φίλο και συνάδελφο, που είχαμε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Μάριο Μάουρο, και ο οποίος για λόγους κατανοητούς εφρόνησε ότι δεν θα έπρεπε να έχει και την θέση ε, του, ε, του ε, Επιτροπής και ε, του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων γιατί αυτή ήταν η θέση στην οποία, ε, ε, κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις μετά από την γενναιόδορη προσφορά του να αποσυρθεί από την Προεδρία του Κοινοβουλίου. Ενδεχομένως και άλλοι μεταξύ ημών μπορεί να ήταν πολύ καλύτερη και ικανότερη από μένα στην ε, κάλυψη των καθηκόντων της θέσεως αυτής. Όμως εγώ ως επιχειρηματία στην αρχή, ως ε, πρόεδρος του Ιταλικού ΣΕΒ αργότερα, ως ε, δήμαρχος του Μιλάνο για εννέα χρόνια και ως βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησα ότι τελικά η πραγματική αιτία ε, της επιτυχίας μου, αν υποθέσουμε ότι επέτυχα σε κάτι στην ε, επαγγελματική μου ζωή, αυτή η αιτία λοιπόν ε, υπήρξε η ποιότητα των καλών μου συνεργατών για τους οποίους πάντα ήμουν ιδιαίτερος υπερήφανος. Και επομένως αναλαμβάνοντας τη θέση αυτή, για την οποία για μία ακόμα φορά σας ευχαριστώ, είμαι βέβαιος ότι θα με στηρίξουν πάντα αυτοί οι συνεργάτες ε, οι οποίοι θα με στηρίξουν γιατί είναι ικανότεροι από μένα και θα είναι σε θέση να καλύψουν ε, την θέση και τις υποχρεώσεις της θέσης. Γι' αυτό λοιπόν αναλαμβάνω την δέσμευση αυτή, την θέση αυτή μάλλον, με μεγάλη ταπεινοφροσύνη, έχοντας πλήρη επίγνωση της δέσμευσης που αναλαμβάνω και που βεβαίως έχοντας κατά νου ότι θα μπορώ να στηριχτώ ε, στα μέλη ε, που τεχνικά με υποστηρίζουν αλλά και όλους τους ε, συναδέλφους που είναι αρμόδιοι για διάφορα θέματα και, τα οποία βεβαίως, και οι οποίοι βεβαίως θα με βοηθήσουν. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη που προβλέπει εκλογή αντιπροέδρων σύμφωνα με ε, τα όσα μου έχουν υποδείξει ε, δεν θα προχωρήσουμε αν αλλά αναπερίπτωση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα να μου γνωστοποιήσει η ομάδα μου την πρόταση για τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Τον λόγο έχει ο εκπρόσωπος της πολιτικής ομάδας. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο για τη θέση του πρώτου ε, αντιπροέδρου, Κύριο Μπέλτερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ε, συγχαρώ εκ βάθους καρδίας ε, για την θέση που μόλις αναλάβατε. Γνωρίζομαι ότι είστε ιδιαίτερος ε, προσφυλής και ε, είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία μας θα είναι ιδιαίτερος καρποφόρα. Θα ήθελα να σας υποβάλω τον κύριο Ρέχα σαν πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι γνώστης των διεθνών θεμάτων Ζητούμε συγγνώμη, έγινε ένα λάθος το όνομα. Ε, είναι... Και γνωρίζομαι από χρόνια την δράση του και την ε, δυνατότητα που είχε να αναπτύξει την πολιτική του δράση από τις θέσεις από τις οποίες πέρασε και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ικανότατο στη θέση του πρώτου αντιπροέδρου. Παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ μπορώ να εκφράσω την θετική μου ψήφο υπέρ αυτής της πρώτης αντιπροεδρίας. Θα ήθελα όμως να προσθέσω μια πολιτική θεώρηση. Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ε, μια πρόταση η οποία πολιτικά αφορά έναν άνθρωπο ε, πολύ ικανό βεβαίως, αλλά που όμως είναι ευρωσκεπτικιστής ε, και εκφράζει αυτήν την ευρωσκεπτικιστή προσκεπτικιστική τάση. Γι' αυτό λοιπόν στο μέλλον νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, δηλαδή ε, θα πρέπει να δεσμευτεί για μια πραγματική εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική και βεβαίως ε, να καλύψει την ε, θέση, αυτός, αυτή τη θέση ο κύριος Προβέρα με ικανότητα και με ευρωπαϊκή διάθεση. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να πάρω το λόγο έτσι ώστε να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα και έτσι ώστε να έχουμε μια πραγματικά φιλοευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Ε, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει και μια άλλη παρέμβαση. Ο κύριος Τάνοκ νομίζω. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώ ήθελα να πάρω το λόγο. Δεν γνωρίζω τον κύριο Προβέρα, τον έχω συναντήσει για πολύ λίγο, αλλά είμαι αντίθετο σε οποιονδήποτε αναφέρεται στο γεγονό ότι είναι ευρωσκεπτικιστή. Είμαστε πραγματιστές και ο αξιότιμος ε, συνάδελφο Γκάλαχ και ο συνάδελφος Βανόρντεν ήταν αντιπρόεδρη αυτή τη Επιτροπής εδώ και χρόνια. Και νομίζω ότι αν υπάρχει κάποιο ευρωσκεπτικιστής, ο κύριος Βανόρντεν είναι ο κατεξοχήν ευρωσκεπτικιστής. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει να, υπάρχει, να χρησιμοποιηθεί αυτό ω φραγμό για να εκλεγεί κάποιος ως πρώτο αντιπρόεδρος τη Επιτροπή, σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Τάνοκ για την παρατηρήσή σας και τώρα έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος, η κυρία συγγνώμη, Λούνατσεκ. Ευχαριστώ <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος των Πρασίνων ε, θέλω και εγώ να πω ότι εμείς ε, θα ψηφίσουμε υπέρ, θα υπερψηφίσουμε για τον κύριο Προβέρα στη θέση του πρώτου αντιπρόεδρου. Όμως επιτρέψτε μου να πω και λίγα λόγια για την ε, αξία και την πολιτική σημασία αυτή τη θέση. Κοιτάξτε, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι στην Ευρώπη να έχουμε μια πολυσχηδή εκπροσώπηση και βεβαίω αυτό αφορά και τις θέσεις των Προέδρων. Άρα δηλαδή οι αντιπρόεδροι τους οποίους ε, καλούμεθα να εκλέξουμε και αυτοί θα πρέπει να εκφράζουν την Ευρώπη της ε, πολυμορφίας, την Ευρώπη όπου γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των ετούντων άσυλο. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ε, Ενωμένη Ευρώπη. Άρα δηλαδή όλα αυτά πρέπει να συνδέονται και με τα αξιώματα που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θεωρώ ότι ο κύριος Προβέρα πράγματι θα παίξει σημαντικό ρόλο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, κυρία Λούνατο, για την παρέμβασή σας. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, παρακαλώ. Ο κύριος Σεβερίνο. Κύριε Πρόεδρε, Βεβαίως, έχουμε ως ε, ένδειξη και ως κατευθυντήρια γραμμή το σύστημα Hunt, ε, το οποίο μας κατευθύνει όσον αφορά τους αριθμούς ε, των πολιτικών ομάδων και τις αντιστοιχίες στους αντιπρόεδρους κτλ. στο σώμα. Και είμαι βέβαιος πως θα τηρηθεί ο κανόνας αυτός. Το πρόβλημα είναι πως οι συνάδελφοί μου έχουν μια πολύ ισχυρή πολιτική επιφύλαξη. Πρόκειται για την επιφύλαξη που εκφράζεται όχι προς τον κύριο Προβέρα, αλλά προς το κόμμα το οποίο αντιπροσωπεύει. Και γι' αυτό και Θέλαμε να κάνουμε αυτή την ξεκάθαρη δήλωση, μια δήλωση ε, επιφύλαξης και ανησυχίας. Μια δήλωση που εκφράζει την επιθυμία ότι αν τελικά ο κύριος Προβέρα εκλεγεί θα μπορεί να υποστηρίξει μια υπερευρωπαϊκή πολιτική και επιλογή. Και έπειτα οι συνάδελφοι, ε, λόγω όλων αυτών που σας ανέφερα, αποφάσισαν αν γίνει ψηφοφορία να απέχουν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κυρία Σεβέριν. Ζήτησε το λόγο ο συνάδελφος Μπροκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για την εκλογή σας και είμαι σίγουρος ότι υπό τη δική σας την καθοδήγηση και με την εμπειρία που διαθέτετε θα περάσουμε δυόμιση χρόνια πολύ ενδιαφέροντα ε, θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστώ και τον κύριο Σάιρους Βόλσκι, ο οποίος ε, νομίζω με ιδιαίτερο επαγγελματισμό και γνώσεις διεύθυνε τις συζητήσεις ε, στην Επιτροπή μας τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω και μία παρατηρήση στη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Κοιτάξτε, εγώ συμμερίζομαι τις ανησυχίες ε, που εξέφρασαν κάποιοι συνάδελφοι όσον αφορά ε, τη στάση ενός ευρωβουλευτού αν είναι φιλοευρωπαϊκή ή ευρωσκεπτιστική, σκεπτικιστική. Απ' την άλλη όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει καμία πολιτική δέσμευση ε, γιατί αλλιώς ε, το παρελθόν θα είχαμε αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Ο κύριος Προβέρα θα είναι αναγκασμένος ε, να υιοθετεί και να εκπροσωπεί τη θέση της Επιτροπής μας. Γιατί αν δεν το κάνει αυτό, τότε καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα. Θα πρέπει όμως να του δώσουμε την ευκαιρία που δικαιούται να εκφράζει την πλειοψηφία της Επιτροπής μας απέναντι στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Γι' αυτό λοιπόν εκ μέρους της δικής μας πολιτικής ομάδας θέλω να σας πω ότι εμείς τηρούμε αυτά που έχουμε συμφωνήσει, τηρούμε τους κανόνες και θα υπερψηφίσουμε τον κύριο Προβέρα. Μάλιστα, έχω την εντύπωση ότι με την παρέμβαση του συναδέλφου Φαν θα μπορέσουμε να κλείσουμε τη συζήτηση και να περάσουμε πίτα στην ε, εκλογή του υποψήφιου αντιπρόεδρου. Φανόρδεν, τελευταία παρέμβαση έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίσης θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας ως πρόεδρο αυτής της Επιτροπής. Απλώς ε, θεωρώ πως ε, θα πρέπει να αντιτεθώ στα σχόλια τα οποία έγιναν. Εγώ δεν ε, φέρω κανένα ε, δαυλό υπέρ του υποψηφίου, αλλά Έχουμε όλοι εκλεγεί με δημοκρατική εντολή από τους εκλογείς μας και πολλοί από τους εκλογείς μας έχουν διαφορετικές απόψεις για τη φύση και τη μελλοντική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι που αντιπροσωπεύουμε. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Και δεν νομίζω πως είναι καθόλου σωστό να προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε οποιαδήποτε είδου ορθοδοξία για την φύση των ανθρώπων που εκλέγονται ω αντιπρόεδροι ή πρόεδροι των επιτροπών. Αντιπροσωπεύουν όλες τις απόψεις, ε, αντιπροσωπεύονται μάλλον όλες οι απόψεις στο Κοινοβούλιο με σωστό και δημοκρατικό τρόπο και σύμφωνα με τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούμε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα όσα λέμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Βαν και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι ή αν κάποιος από τους ε, παρόντες που αντιπροσωπεύουν ε, που αντιπροσωπεύει μάλλον το απαραίτητο ποσοστό να ζητήσει, θέλει να ζητήσει μυστική ψηφοφορία. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε δηλώνουμε ότι εκλέγεται διαβοή ο κύριος Προβέρα ως πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τον καλό να καθίσει δίπλα μου. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στην εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια απέφχομαι μια τέτοια μακρά συζήτηση, αλλά εάν συμβεί θα το δεχτώ. Λοιπόν, θέλει κάποιος να παρουσιάσει τον δεύτερο υποψήφιο αντιπρόεδρο. Κύριε Σεβερίν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, διότι ξέχασα στην προηγούμενη μου παρέμβαση να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στην θέση αυτή και να εκφράσω την ελπίδα μου και την επιθυμία μου να συνεργαστούμε μαζί σας ε, αρμονικά για το καλό του σώματος και των πολιτών μας. Τώρα, όσον αφορά την πρότασή μας για το δεύτερο αντιπρόεδρο, της Επιτροπής Εξωτερικών είναι ο κύριος Ιωάννης Σαπάσκου που είναι γνωστός από τα πιο όρημα μέλη γιατί δεν είναι ε, όλοι ε, ε, παλιά, παλιά μέλη. Οι περισσότεροι θα το γνωρίζουν από την προηγούμενη ε, θητεία. Ήταν τέταρτος αντιπρόεδρος στην προηγούμενη θητεία και τώρα ελαφρώς προάγεται, αν τον ψηφίσετε βέβαια, ως δεύτερος αντιπρόεδρος. Νομίζω πως είναι αρκετά πεπειραμένος σε αυτήν την θέση. Επίσης διατέλεσε Υπουργός Αμήνης της Ρουμανίας πριν από λίγα χρόνια. Είναι λοιπόν πεπειραμένος στις διεθνείς σχέσεις και νομίζω πως με τη δική του συμβολή θα έχουμε μεγάλη προστιθέμενη αξία στη δουλειά μας. Ευχαριστούμε κύριε Σεβερίν και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα ε, ρωτήσω εάν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι και αν κάποιος από τους παρόντες, ο οποίος να εκπροσωπεί το αντίστοιχο ποσοστό που προβλέπεται από τον κανονισμό, θέλει να προτείνει μυστική ψηφοφορία για τον δεύτερο αντιπρόεδρο. Νομίζω πως ε, όχι. Οπότε σας καλώ αφού κηρύξουμε την εκλογή του διαβοής θα καλέσω τον κύριο Πασκούν να έρθει στο έδρανο της Προεδρίας. Προχωρούμε τώρα στην ε, εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Τον λόγο έχει ο εκπρόσωπος του κόμματος που δικαιούται την τρίτη αντιπροεδρία. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Μπροκ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εκ μέρου ε, του συναδέλφου Σαλαφράγκα και του ΕΛΚ ε, θα ήθελα να σας προτείνω Ντομινίκ Μποντής για αυτή τη θέση. Μισό λεπτό. Α, ε, Λοιπόν, δεν έχει καμία σχέση αυτή η παρατήρηση που έγινε εκτό μικροφόνου. Επανέρχεται ο μιλητή. Ντομινίκ Μποντή. Ε, Μια πεπειραμένη συνάδελφο ε, που ε, ναι μεν τώρα ήρθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά για πολλά χρόνια ήταν ε, ε, δήμαρχος ε, της Τουλούζης έχει συγκεντρώσει μεγάλη εμπειρία και θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να στηρίξουν την πρότασή μας. Eh, Εάν κανείς από τους ε, παρόντες ε, δεν προτείνει μυστική ψηφοφορία και αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι όπως ε, νομίζω μπορούμε λοιπόν να εκλέξουμε διαβοή στον κύριο Ντομινίκ Μποντίσε για την θέση του τρίτου αντιπροέδρου και τον καλό να καθίσει και αυτός στο έδρανο της Προεδρίας. Προχωρούμε τώρα στην εκλογή του τετάρτου αντιπροέδρου πάντα με τον ίδιο τρόπο. Καλό λοιπόν τον ε, συνάδελφο ο οποίος ε, έχει αναλάβει το ρόλο αυτό να υποβάλει την υποψηφιότητα του τετάρτου αντιπροέδρου. Ποιος έχει το λόγο? Ο κ. Μέγερ. Καταρχήν θα ήθελα εξ ονόματος της ε, ΓΚΟΕ, της ομάδας μας, Θα ήθελα, λέω, να σας συγχαρώ για την, το διορισμό σας. Θα ήθελα να προτείνω τον κύριο Μελενσόν στη, για τη θέση του, του τετάρτου αντιπρόεδρου. Έχει μακρά ε, ε, νομοθετική εμπειρία για 20 χρόνια στην Γαλλική Γερουσία και ήταν και γραμματέας της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μέγερ. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, υπάρχει κάποια άλλη υποψηφιότητα. Ε, ζητά κανείς μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του τετάρτου αντιπροέδρου. Αρνητική απάντηση και στα δύο ερωτήματα. Και επομένως κηρύσσεται εκλεχθής διαβοής στην θέση του τετάρτου αντιπροέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κύριος Μελενσόν και τον παρακαλώ να έρθει να καθίσει στο έδρανο της Προεδρίας.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 ε, αγγελίες που αφορούν και ανακοινώσεις που αφορούν τις ε, προσεχείς μας εργασίες. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, όπως ε, ήθιστε να συμβαίνει όταν βρισκόμαστε απέναντι σε ιδιαίτερες δεσμεύσεις, να γυρίσουμε λίγο σε το παρελθόν μας, γιατί αυτό ήθιστε να κάνουμε. Γυρνούμε στις ρίζες μας όταν βρισκόμαστε απέναντι σε μελλοντικά σημαντικά πράγματα. Και από τη στιγμή που έχουμε και εδώ ε, πολλούς εκπροσώπους που έχουν ασχοληθεί με τις πόλεις, θα ήθελα να σας ε, αναφέρω μία φράση του Αγίου Αμβροσίου, του προστάτη του Μιλάνο, που ίσως ε, πολλοί γνωρίζετε ότι δεν γεννήθηκε στο Μιλάνο, αλλά στη Γερμανία, στο Τρίερ. Άρα είναι ένας Ευρωπαίος προστάτης. Όταν οι τυχαίες συνθήκες και τα τυχαία περιστατικά και ε, όπως συμβαίνει και αυτή τη στιγμή σε μένα και δεν θέλω να είμαι ε, προσβλητικός. Όταν λοιπόν εκείνος έγινε επίσκοπος, ξεπερνώντας μια σειρά από προβλήματα, άρχισε να διδάσκει αυτά που έπρεπε εκείνος να μάθει. Με όσο χιούμορ λοιπόν διαθέτω, γιατί βεβαίως είναι εκτός αναλογιών αυτή η σύγκριση, μπορώ να πω ότι εγώ αναλαμβάνω το ρόλο του Προέδρου με αυτό το πνεύμα, γνωρίζοντας δηλαδή ότι ε, θα έχω δίπλα μου εξαιρετικούς ανθρώπους με περγαμινές σημαντικές και επομένως μια σειρά, μια ομάδα μάλλον από συνεργάτες που θα με στηρίξουν με μεγάλη αξιοπρέπεια και που, από τους οποίους έχω πάρα πολλά να μάθω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για την προσοχή που δείξατε, για τον πολύ ευγενή και ορθό τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η συνεδρίαση αυτή. Ξεκινήσαμε ε, με την ε, ορθή ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων που εξεφράστησαν όμως ε, με τάξη και ευγένεια. Να πω ότι την επόμενη εβδομάδα, 3η 21 Ιουλίου και στις 3 το απόγευμα ή στην αίθουσα Γιάν 2Q2 θα λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίασή μας. Κυρία Μπράνερ, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ κυρία Μπράνερ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ όλους για την εκλογή σας. Εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων θα ήθελα να πω ότι είναι κρίμα που δεν υπάρχει ούτε μία γυναίκα στο Προεδρείο της Επιτροπής μας. Είναι πράγματι πολύ λυπηρό. Σας εύχομαι όμως καλή επιτυχία και αναμένω καλή συνεργασία μαζί σας και ε, Συμμερίζομαι απόλυτα το σχόλιο σας και το ενστερνίζομαι. Όμως, θα ήθελα να προσθέσω ότι έστω και αν οι γυναίκες δεν είναι στο Προεδρείο, υπάρχει σημαντική αντιπροσώπευση γυναικών στους συντονιστές που κατά κάποιο τρόπο αντισταθμίζει στην ηγεσία ας πούμε της, ε, ε, της Επιτροπής μας αυτό το άλλο μισό του ουρανού. Να σας πω επίσης ότι θα έχουμε διευρυμένο προεδρείο από τις 11.30 μέχρι τις 12.30 στην αίθουσα ΑΣΠ 1Ε1 στις Βρυξέλλες την ίδια μέρα, 21 Εβδόμου δηλαδή. Θα έχετε βεβαίως και την απαραίτητη γραπτή πληροφόρηση. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Ε, εύχομαι σε εσά και στον εαυτό μου βεβαίως ε, ε, ευόδος των εργασιών μας.